παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη. Ένα εκατομμύριο Ιγουροί κρατούνται σε στρατόπεδα φυλακές υψηλής ασφαλείας. Ε, υπάρχει μία προσπάθεια αλλαγής πεπιθήσεων ε, όμως αυτά τα στρατόπεδα είναι και σε συνεχή παρακολούθηση. Δεν είναι μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Είναι ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δεν αρκούν οι δημόσιες δηλώσεις. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με την Κίνα. Να γίνει μια έρευνα στις ευρωπαϊκές εταιρείες που δρούν στη Σινγκιάνγκ. Είπατε εκπρόσωπε, εσείς και η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μιλήσατε για το πώς η Κομισιόν είναι μια γεωπολιτική επιτροπή. Θα παραμείνει λοιπόν σιωπηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα αναλάβει σοβαρή δράση κατά της Κίνας. Επιπλέον, ποια είναι η στρατηγική που θα διασφαλίσει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις απειλές κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πηγαίνουν, ε, που χρησιμοποιεί η Κίνα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και συλλογής ε, δεδομένων, χωρίς διαφάνεια για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο, ε, Πέτρα Αστρεπίτσιους, έχετε ένα λεπτό. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, συνάδελφοι, η παγκόσμια δύναμη της Κίνας ε, χτίζεται πάνω στην καταστολή και το βάσανα του λαού τη. Υπήρξε δηλώσει ε, για λήψη, παράνομη λήψη οργάνων στην Κίνα. Έχουμε ένα πονίδι στο σύστημα. Αυτά τα στρατόπεδα αναμόρφωσης που δεν περιορίζονται στην ε, πολιτιστική αφομοίωση των Ουιγούρων. Είναι ένα μαζικό πρόγραμμα εκπαίδευση στο χώρο εργασία, όπως το λένε για να έχουν φθηνά εργατικά χέρια τα κινέζικα εργοστάσια που είναι κομμάτι της παγκόσμιας ε, αλυσίδας παραγωγής. Οι πολιτικές ελευθερίες των πολιτών της Κίνας δεν γίνονται σεβαστές. Η πολιτιστική αφομοίωση δεν είναι το δόγμα και όχι η πολιτιστική ε, ποικιλομορφία. Η παγκόσμια, ε, ε, το Παγκόσμιο Νόμος Μακνίσκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικότερος Νόμος Μακνίσκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια λύση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επίσης θα εμπόδιζε και άλλες χώρες από το να, να παραβιάζουν τα δικαιώματα και να κάνουν παρόμοια εγκλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σόιντροβα έχει τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, η Κίνα και όσα γίνονται στην περιοχή της Ξινιάνγκ, η παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη χρήση τεχνολογικών μέσων ή υπερσύγχρονων για την παρακολούθηση των πολιτών είναι απαράδεκτα. Με το, το Κοινοβούλιο ε, προσπαθήσαμε να στείλουμε ένα χειρότατο μήνυμα με την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στον κύριο Τότη. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή του και την απελευθέρωση όλων των εκατοντάδων χιλιάδων κρατουμένων. Θέλουμε να ε, να απελευθερωθεί και ο πρώην κυβερνήτη τη περιοχή, ο οποίο απελείται με θανατική καταδίκη, με την εκτέλεσή του. Η κόρη του Ιλχάμ μα είπε ότι φοβάται. Φοβάται και το γεγονό ότι. Ε, το κοινοβούλιο τον βράβευσε, μπορεί να απειλεί ακόμη περισσότερο τη ζωή του. Η κυβέρνηση της Κίνας είναι υπεύθυνη για μια πολιτιστική γενοκτονία στην περιοχή της Ξινγιάν και χρειάζονται εδώ στοχευμένες κυρώσεις. είπατε εκπρόσωπε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας σημειώστε την έκκλησή μας μια νέα στρατηγική για την Κίνα. Μια στρατηγική που πρέπει να χαράξουμε για το μέλλον ζητώντας συγκεκριμένα βήματα πρόοδου για τα θεμελιώδη δικαιώματα από τις κοινωνικές αρχές. Ευχαριστούμε Γιόντσεβα για ένα λεπτό. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα κατάφορες από τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας με τη μαζική παρακολούθηση και εγκλισμό ε, άνω ε, ε του ενός εκατομμυρίου Ουιγούρων και άλλων εθνικών μειονοτήτων στην Κίνα από την αυτόνομη περιφέρεια Ξιν Γιάνκο Ιγούρ κατά την περίοδο του ε, ολοκληρωτισμού και η δική μου χώρα, η Βουλγαρία, πέρασε δύσκολες στιγμές με μια εθνική μειονότητα ε, όπου είδε τα δικαιώματά της να περιορίζονται. Ήταν δύσκολα χρόνια, πέτρινα τα χρόνια εκείνα. Σήμερα η Βουλγαρία είναι παράδειγμα προς μίμηση ε, για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στην εθνική και θρησκευτική της μειονότητα. Ελπίζω η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας που είναι σπουδαία χώρα με αρχές παραδόσεις και πολιτισμό να βρει το δρόμο της προς την προστασία ε, και την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων, όλων των εθνικών ε, μειονοτήτων και να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι παρατηρητές και δημοσιογράφοι να μεταβούν στην αυτόνομη περιφέρεια Ξιν Γιάκ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε, είπατε εκπρόσωπε. Ε, ενώ εμείς ξέρουμε αυτή τη συζήτηση, απευθυνόμαστε στην ουσία στην Κίνα. Το ίδιο σχέδιο για το ψήφισμά μας. Ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαρκώς προασπίζονται τις θρησκευτικέ μειονότητες. Ακόμα και εάν μιλάμε για μια χώρα όπως η Κίνα, το ψήφισμα μας είναι σωστά εξισορροπημένο και πραγματικά εκτιμούμε Ε, το όσο θετικά συμβαίνουν στην Κίνα. 700 εκατομμύρια ε, άνθρωποι βγήκαν από συνθήκε φτώχεια. Υπάρχουν σοβαρέ ε, επενδύσει στι υποδομέ και εγκαταστάσει. Όμω αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το ψήφισμα αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνει στοιχεία. Αναντήρητα γεγονότα τα οποία έχουν επαληθευτεί, τα έχουμε ελέγξει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει θετική απόκριση από την κινέζικη πλευρά. Εάν όμως χρειαστεί, μπορεί να ε, σκίσουμε να προβλέψουμε κυρώσεις για τις εμπορικές μας σχέσεις. Θα πρέπει επιτέλους να κυρώσουν την ε, παγκόσμια συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν ε, ε, υπογράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε και τώρα ξεκινούμε τη διαδικασία Catch the Eye προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου. Ξεκινάμε τον κύριο Χάιζερ, είχατε ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, εδώ η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα, μια μεγάλη δύναμη με ιστορία ιστορία χιλιετίας, χιλιετιών ε, και μεγάλος εμπορικός μας εταίρος. Εδώ όμως δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε στις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Ιδίως στην ε, περιοχή του, της Ξινιάνγκ. Ε, είναι, είναι ένα εκατομμύριο περίπου οι που βρίσκονται σε στρατόπεδα όπως ονομάζονται αναμόρφωσης ενώ είναι συγκέντρωσης, Στατόπεδα συγκέντρωσης είναι. Δεν πάει και ο κόσμος ή και ο θελός. Εδώ λοιπόν αυτό δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Ε, οφείλουμε να οργανώσουμε διάλογο με τους Κινέζους ηθήνοντες και να τονίσουμε ότι αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αντί να προβλέψουμε όμως κυρώσεις, νομίζω ότι ο στόχος ε, ε, πρόσβασης στη χώρα, στην Ξινγκιάν, από διεθνείς, από διεθνείς παρατηρητές και δημοσιογράφους είναι σημαντικό. Εάν δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, εντάξει, αλλά αν διαπιστωθούν συστηματικές παραβιάσεις, τότε οι κυρώσεις θα είναι το μόνο μπορεί να συμβεί. Ευχαριστούμε. Ε, και τώρα κυρία Γουόρντ για ένα λεπτό. Ε, τα κυβερνητικά έγγραφα που διέρευσαν έχουν προσελκύσει την προσοχή στα όσα κάνει η κοινωνική κυβέρνηση στι παραβιάσει ε, δικαιωμάτων των Ιγούρων και άλλων μειονοτήτων. Αυτά που είχαν ξεκινήσει με τη φυλάξη του επικεφαλή του το 2014. Η Κίνα αρνείται τι επικρίσει κατά τη υποβάθμιση των δικαιωμάτων, όμω είναι ένα εκατομμύριο Ουιγούροι, Καζάκοι και άλλοι που πηγαίνουν στα στατόπεδα ε, αναμόρφωση, ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για προσελητισμό πολιτιστικό και πολιτικό. Η Κίνα τα βασανιστήρια αυτά τα αρνείται και μιλά για κέντρα επαγγελματική εκπαίδευση. Λε και πάει να δώσει επαγγελματικέ δεξιότητε σε φοιτητέ. Ε, τα έγγραφα διέρευσαν από, από κυβερνητικού εκπροσώπου που τιμωρούν τα παιδιά φυλακισμένων γονιών και ε, είναι εκείνοι που λαμβάνουν την υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση εντό εισαγωγικών για να μην μπορούν βέβαια να κάνουν τη ριζοσπαστική τρομοκρατική τους δράση όπως έχει χαρακτηριστεί. Είναι εκατοντάδε οι τοπικοί εξωματούχοι που έχουν φυλακιστεί. Ένα φυλακίστηκε γιατί προσπάθησε να σταματήσει τι αυθαίρετε συλλήψει. Εγώ είμαι υπερήφανη που ε, ε, ηγούμε μια εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση που οργανώνει μηνιαίε διαμαρτυρίε, κάθε μήνα διαμαρτυρίε διαμαρτυρίες έξω την ε, πρεσβεία της Κίνας στο Λονδίνο και που ζητά το ε, κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ε, ο κύριος Βουάλλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κίνα, Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη, Αμερική, όπου και αν είναι, καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι φιλελεύθεροι όμως ε, ε, πολιτικοί μιλάνε για τους μουσουλμάνους ενώ στην ουσία έχουν γεωπολιτικούς λόγους. Έχουμε εκατομμύρια μουσουλμάνους που καταδικάζονται και καταλείπονται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή οι χριστιανοί στη Συρία διώκονται. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο ως όπλο για το να υποσκαφτούν συγκεκριμένα κράτη δεν είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Η πρωτοβουλία Belt and Road είναι η ουσία. Το Σινγκιάνγκ ε, βρίσκεται σε αυτό το δρόμο. Γι' αυτό έχει κερδίσει και την προσοχή των Αμερικανών θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή γιατί δεν θέλουν αυτή η πρωτοβουλία που οι Κινέζοι τόσο καιρό ε, σχεδιάζουν να ε, πραγματοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα η κυρία Ντάλη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Daily. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για το China Cables, τα οποία ε, έχουν να κάνουν και με τις τα εκρηκτικά Wikileaks του 2010. Ήταν ένας νέος, ε, μια νέα δημοσιογραφική πρακτική που ε, γύρει το ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν τις κυβερνήσεις. Εδώ έχουμε μια πηγή που υποτίθεται ότι έρχεται από την κινέζικη κυβέρνηση και διαρρέει ένα εγγραφό στα αγγλικά και όχι στα κινέζικα, σε αμερικανικό κοινό ε, που δημοσιεύεται ε, από έναν ε, αμερικανικό μικιό, από μια αμερικανική μικιό που παίρνει και κονδύλια από την Αμερική. Είναι σαν να μας λένε από το Ιράν τι κάνει η Ιρανική κυβέρνηση. Και ας θυμόμαστε, ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να βασιστούμε στους Κινέζους και να κάνουμε πόλεμο με το Ιράν. Και αυτή τη στιγμή μιλά για τις διώξεις των μουσουλμάνων στην Κίνα. Δεν αμφιβάλλω ότι γίνονται τέτοιες διώξεις και το καταδικάζω απερίφραστα. Όμως πολλά κράτη έχουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς ε, που διώκονται. Πού είναι οι καταγγελίες γι' αυτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ χρησιμοποιούνται για γεωπολιτικούς λόγους. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλοι αγορητές. Τώρα δίνω το λόγο στον είπα το εκπρόσωπο. Ζωζεφ Μπορέλ. Ε, Ζωζεφ Μπορέλ Φοντέλες, έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ε, καταλήγω ότι η πλειοψηφία, για να μην πω ομοφόνος, το σώμα ανησυχεί για την κατάσταση στην Κίνα και ζητά από την Κίνα να αλλάξει δραστικά τις πολιτικές της στην περιοχή αυτή. Ειδικά την χρήση των ε, στρατοπέδων πολιτικής αναμόρφωσης ε, και τις τεχνικές μαζικής παρακολούθησης. Αυτά λέγονται ε, ότι γίνονται για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Όμως πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι δίνετε προσοχή σε αυτά τα θέματα και ότι υποστηρίζετε αυτό το ζήτημα, το βάζετε ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, σας θαυμάζω γιατί αλήθεια η ε, ενεργά προωθεί αυτό το αφήγημα της ε, πάταξης του ιστρομοκρατίας ε, στη Σινγκιάνγκ και παίρνει μεγάλη υποστήριξη από πολλές χώρες. Η διάσκεψη Λάμπη, ας πούμε, είναι τα μέλη της που υποστηρίζουν, για να μην πω για τη Γενική Συνέλευση, μια ομάδα 22 χωρών πολλά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη μεταξύ αυτών έκαναν μια κοινή δήλωση την στις, ε, για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Ιγούρων. Την ίδια στιγμή είχαμε 54 χώρες ε, με ε, την Λευκορωσία στο, στην κεφαλή να λένε ότι η Κίνα κάνει καλά που κάνει δράσεις κατά της τρομοκρατίας. Φαίνονται λοιπόν ότι η διεθνής κοινότητα δεν είναι ομόφωνη. Εμείς οι Ευρωπαίοι Πρέπει λοιπόν να είμαστε αφοσιωμένοι ε, και μπορούμε να πούμε ότι ε, είμαστε ισχυροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέραμε τις ανησυχίες μας για τη Σινγιάνγκ με ξεκάθαρο τρόπο, όπως και τη χρήση των μαζικών παρακολουθήσεων. Έχουμε κανόνες ε, για την ε, παρακολούθηση και τους ελέγχους των προϊόντων διπλής ε, χρήσης. Παρακολουθούμε τις βασικές τεχνολογίες και τα ελέγχουμε για λόγους ασφαλείας. Και βεβαίως έχουμε ακούσει για την καταναγκαστική εργασία από το 2018. Όταν ξεκινήσαμε τον διάλογο μας με την Κίνα και σε κάθε διμερή συνάντηση με αυτούς. Είπαμε λοιπόν στις εταιρείε μας ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ε, πρέπει να ε, διατρέχει όλη τους την ε, αλυσίδα τροφοδοσίας. Οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν ιδιαίτερα ως προς την επιβολή κυρώσεων στην Κίνα. 28 κυβερνητικά όργανα και εταιρείε στη Σινγκιάνγκ υπέστησαν κυρώσεις. Εμείς δεν το κάναμε, είχαμε άλλο σύστημα. Ξέρετε ότι προσπαθώ να το βελτιώσω ξεκινώντας αυτή την πρωτοβουλία που θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει να εγκρίνουμε κάτι παρόμοιο με τον νόμο Μανίτσκι. Θα σας ε, ενημερώσουμε, ε, σας ενημερώσαμε για τη δουλειά που ήδη ξεκίνησε. Χρειάζομαι όμως ομοφωνία στο Συμβούλιο για να κάνω κάτι τέτοιο. Και θα παλέψω γι' αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε δυνατοί αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και τον διάλογο. Ο διάλογος δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και οι δύο τρόποι μπορούν να ακολουθηθούν. Χρειαζόμαστε όμως και την ισχυρή δέσμευση και εμπλοκή και δράση ε, σε αυτό το θέμα να τη συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, Έχω λάβει πέντε προτάσεις, πέντε σχέδια ψηφίσματος για τη συζήτηση αυτή. Η συζήτηση λίγη και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα να προχωρήσουμε, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δήλωση του του εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής για την ε, κατάσταση στην Βενεζουέλα και την, μετανάστευ... την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Σε ό,τι αφορά το AI και την γαλάζια κάρτα, μπορείτε είτε ηλεκτρονικά είτε ο συνήθω να ε, ζητήσετε το λόγο. Οι οδηγίες υπάρχουν στο έγγραφο στην του της αίθουσας. Και τώρα ο λόγο στον ύπατο εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ζωζέ Μπορέλ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη πολιτικό αδιέξοδο και δεινή οικονομική κατάσταση επικρατεί στη Βενεζουέλα με ολέθριο αντίκτυπο στη χώρα. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Πάνω από 21% του πληθυσμού υποφέρει από υποσυτισμό. 25% επιβιώνουν από ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μπορούσα να προσθέσω πολλά αριθμητικά στοιχεία, τα περισσότερα τα γνωρίζετε. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η κρίση. Το 70% των παιδιών δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχειώδη, φάρμακα, νερό, ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Καράκας ε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά ε, περισσότερες περιοχές της χώρας ε, υποφέρουν από συχνές τακτικές διακοπές ρεύματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μόνιμη παρουσία στη χώρα εγκαθιδρύσει για να παρακολουθεί καλύτερα την κατάσταση. Πάνω από 170 εκατομμύρια έχουμε δώσει από το 2018 και περίπου 320 εκατομμύρια μαζί με τη βοήθεια των κρατών μελών και ε, εντός της Βενεζουέλας αλλά και στις γειτονικές χώρες. Γύρω στα δύο τρίτα της άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν δοθεί σε δράσεις εντός της Βενεζουέλας και είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί και το υπόλοιπο τρίτο πηγαίνει στις γειτονικές χώρες. Ε, επειδή δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες δράσης εντός της χώρας, Υπάρχει μια διεθνή ομάδα επαφών με ανθρωπιστική διπλωματία και προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρξει ένας χώρος ε, όπου να μπορούν να δρουν οι ανθρωπιστικοί ε, παράγοντες εκεί. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, ε, το σημαντικότερο μεταναστευτικό κύμα στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία. Κάθε χώρα, πάνω από 5.000 πολίτες της Βενεζουέλας φεύγουν από τη χώρα, ήδη έχουν φύγει 5 εκατομμύρια. Στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική έχει αυξηθεί η διασπορά. Είναι περίπου 4 εκατομμύρια οι Βενεζουελάνοι αυτή τη στιγμή. Ε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι ε, αναμένεται να αυξηθούν αυτά τα νούμερα μέχρι τα 4 εκατομμύρια επιπλέον και να φτάσει 5 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη του έτους, του επόμενου έτους. Θα ήθελα να επενέσω τις χώρες της περιοχής για τις αξιέπαινες προσπάθειές τους για να βοηθούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, αλλά συνολικά χρειάζεται ε, βοήθεια όλο και περισσότερη. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, έχουν ένα ε, σχέδιο για περιφερειακή απάντηση ε, που αντανακλά τις ανάγκες χρηματοδότησης που έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με την περσινή περίοδο και έχουν φτάσει περίπου τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αριθμοί είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ε, ότι και κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να αρνούνται αυτές τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές. θα πρέπει ε, να διατηρηθεί αυτή η ε, προσοχή η διεθνής που δημιουργήθηκε ε, τον Οκτώβριο με τη διεθνή διάσκεψη που διοργανώσαμε στις Βρυξέλλες δεν στριμώχθηκαν οι δωρητέ εκεί. Θα πρέπει να διοργανώσουμε και άλλη διάσκεψη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ό,τι και να κάνουμε πάντω, και ε, όσο βαθιά και αν σκάψουμε ε, στο κορβανά της αλληλεγγύης μας, δεν φτάνουν ποτέ τα χρήματα που έχουμε για να αντιμετωπιστεί τέτοια τεράστια κρίση. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να δίνουμε τροφή σε εκατομμύρια ανθρώπων. Η Βενιζουέλα παραμένει πλούσια χώρα. Και παρά το γεγονός ότι είναι βαθιά η φτώχεια, ε, στην οποία έχει ρίξει το λαό της, έχει από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικών πόρων. Επίσης έχει και σημαντικά ε, ε, στοιχεία περιουσιακά και πολλά από αυτά είναι στο εξωτερικό. Σίγουρα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν για να ανακουφιστεί ο πόνος και τα δυνά των πολιτών της χώρας Γιατί η αλληλεγγύη δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Είναι τεράστιες ανάγκες και πολλοί άνθρωποι. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε δημιουργικές λύσεις για να κινητοποιήσουμε κάθε είδους πόρο ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια κρίση. Και ελπίζω ή στο προσεχές μέλλον να μας απασχολήσει αυτό και να βρούμε νέες ιδέες. Πάντως, κάπως πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο και το πολιτικό αδιέξοδο που επικρατεί και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Για τα καλά. Είναι η πολιτική κατάσταση. Και τέλος, να είμαι σαφής, η μόνη μακροπρόθεσμη λύση στην ε, πολυδιάστατη κρίση της Βενεζουέλας μπορεί μόνο μετευθεί μέσω μιας ε, δημοκρατικής διαδικασίας στη Βενεζουέλα που θα οδηγήσει σε ελεύθερες προεδρικές εκλογές. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε για την πολιτική λύση για να αντιμετωπίσουμε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις από τη μεταναστευτική σκοπιά και από τη σκοπιά της ευημερία των λαών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ θα δώσω το λόγο στο Λεοπόλντο Λόπες Χίλ για δύο λεπτά. Το είπε μόλις ο ύπατος εκπρόσωπος, η μετανάστευση στη Βενεζουέλα έχει λύσει είναι η έξοδος από αυτό το καθεστώς και η επιστροφή στη δημοκρατία. Τα μπλοκάμπια του Νικολάς Μαδούρο και πάλι θέλουν να εξαλείψουν οποιαδήποτε νόμιμη εξουσία στη Βενεζουέλα, την Εθνοσυνέλευση. Τις τελευταίες ώρες ε, πολλοί βουλευτέ κατηγορήθηκαν και διώχθηκαν παράνομα, εξορίχθηκαν ε, και τους αφαιρέθηκε η ασυλία τους για να αποφύγουν ε, Χουάν Γκουαϊντό που αναγνωρίζεται από αυτό το κοινοβούλιο και η Εθνοσυνέλευση να συνεχίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία. Είναι ντροπιαστικό να ε, βλέπουμε ε, ότι καταστέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και ο οργανισμός αυτός ουσιαστικά μετατρέπεται σε κάποιους τυράννους που η κυρία Μπατσελέ καταγγέλει την συνέχιση των καταχρήσεων. Η έλλειψη σεβασμού της αξιοπρέπειας του λαού έχει προκαλέσει μια μετανάστευση 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το 20% έχει εγκαταλείψει τις αιστείε του Ένα στους 10, ένα στους 5 διορθώνει ο κατοίκου. 300.000 Βενεζολάνου έχουμε σήμερα στην Ισπανία. Και ε, είναι πρώτη ε, στο αιτήσει ασύλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση και να θέσει τέλο στη δικτατορία με κατάλληλη ηγεσία από τον είπα το εκπρόσωπο και με την επιβολή κυρώσεων ε, όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και λυπάμαι που ε, όπως ε, είπε σήμερα το πρωί και η εφημερίδα ε, El Mundo, λυπάμαι ότι που μόνο ο Μαδούρο ή ο Τραμπ κατηγορούνται για το τι σημαίνει στη Βενεζουέλα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Χαβιλόπες, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον είπα το εκπρόσωπο, τον ε, κύριο Γιωσέ Μπορέλ. Ε, μιλάμε για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, τα δεινά που υφίσταται η Βενεζουλάνη και το τεράστιο αντίκτυπο που έχει στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής. Ε, και θα ήθελα να δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για το τι βιώνεται σήμερα στη Βενεζουέλα. Το 82% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο γορό. το 53% ε, υφίσταται περικοπές στις προμήθειες και έχουμε έλλειψη στα φάρμακα. 11 εκατομμύρια Βενεζολάνοι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Μεταξύ αυτών, πολλοί εκτός της χώρας, το 80% στην περιφέρεια στη Λατινική Αμερική των εκτοπισμένων και 35% του συνόλου του πληθυσμού. Γι' αυτό μιλάμε για μια μαζική έξοδο πρωτοφανή στην ε, περιοχή, 4,5 ε, εκατομμύρια άτομα με τεράστιο αντίκτυπο, όπως υπόθηκε εδώ, σε ένα μακρύ κατάλογο χωρών, Κολομβία, Περού, Αργεντινή, Χιλή, που επίσης πρέπει να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια, όταν ε, ήδη έχουν ε, πολύ σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν δράση και κυρίω να υπάρξει οικονομική υποστήριξη σε μια τέτοια κρίση. Τα Ηνωμένα Έθνη ε, έκανε μια αξιολόγηση στα δύο δισεκατομμύρια τι ανάγκε των Βενεζολάνων εντό και εκτό τη χώρα φέτο. Μόνο το 25% μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε αυτού του αριθμού. Γι' αυτό ζητάμε μια δημοκρατική έξοδο για τη χώρα, όπως ε, έγινε το προηγούμενο ε, ο από την κυρία Μεογκερίνη να υπάρξει προβολή του τι συμβαίνει με τους μετανάστες ε, στη Βενεζουέλα και θέλουμε πρωτοβουλίες όπως είναι το πετρέλαιο αντιτροφίμων και επίσης να υπάρξουν ε, ε, κάποιες κυρώσεις. Όμως ε, πρέπει να προσέχουμε οι κυρώσεις να μην θίγουν τον πληθυσμό γιατί ήδη τιμωρούνται αρκετά οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας Renew, η κυρία Χαράντσοβα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ τον είπα το εκπρόσωπο. 4 εκατομμύρια Βενεζολάνοι δεν ε, είχαν άλλη λύση παρά να φύγουν από τη χώρα τους. Οι εκτιμήσεις για το 2020 είναι τόσο υψηλές όπως τα 8 εκατομμύρια, πολύ πιο πάνω από τους εκτοπισμένους στη Συρία. Η διαφορά μεταξύ των δύο, η Συρία είναι μια χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, η Βενεζουέλα όχι. Όμως ε, οι συνθήκες ε, που υφίστανται καθημερινά οι Βενεζολάνοι δεν διαφέρουν πάρα πολύ από μια περιοχή εμπόλεμης σύραξης. Αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα είναι μια τραγωδία και πολύ περισσότερο επειδή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση ήταν το αποτέλεσμα των πολιτικών του καθεστώτος ε, και της, του δισταγμού του να παραδεκτεί την ύπαρξη του προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει κάθε υποστήριξη που μπορεί για να ανακουφίσει την ανθρωπιστική, η ανθρωπιστική κρίση. Όμως αν δεν επιληθεί σε εσωτερικό επίπεδο η πολιτική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση δεν θα έχει τέλος. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βενεζουέλα θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η εξή, να σκείται πίεση στο καθεστώς του Μαδούρο προκειμένου να κάτσει και να διαπραγματευτεί μια ειρηνική μετάβαση. Όπως ε, έχω πει ε, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να γίνει είναι οι επιλεκτικές κυρώσεις ε, κατά αξιωματούχων του καθεστώτος και γι' αυτό θα πρέπει να διευρύνουμε τον κατάλογο των επιλεκτικών κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων, Αλής Κούνκε. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιωσέπ Μπουρέλ. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να θίξετε αυτό το πολύ δύσκολο και σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάνθρωπη κατάσταση που συνεχίζεται τόσοι και τόσοι έχουν φύγει από τη χώρα, υπάρχουν ε, ταραχές, βία, πείνα. Και θέλω να επισημάνω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν φύγει από τη χώρα, ψάχνοντας να βρουν καταφύγιο σε γειτονικέ χώρες. Νομίζω ότι αυτό καθιστά προφανές ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία τελικά δεν λύνονται. Ούτε υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πλέον αντίκτυπο και σε άλλες χώρες ε, ε, στην ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα η κατάσταση όλο ένα και χειροτερεύει. Τον Οκτώβριο, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τι γειτονικέ χώρε στη Βενεζουέλα να δείξουν αλληλεγγύη προ ε, τη γείτονά του. Και εμεί ω πράσινοι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αλληλεγγύη ε, θα είναι κάτι το οποίο θα δείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε να δράξουμε την ευκαιρία να δείξουμε πραγματικά την αλληλεγγύη μας, γιατί μέχρι τώρα μόνο λόγια έχουμε ακούσει. Έχουμε πει ότι θα ε, αντισταθούμε στους ε, διεφθαρμένους που καταπιέζουν τον κόσμο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας ID, ο κύριος Μαριανή, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η διπλωματία είναι πλήρως ξένη προς ε, τις ε, φιλοσοφικές ε, προεκτάσεις που χρησιμοποιούνται εδώ και όλη η πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι, και η στάση της απέναντι στην Αμερική δείχνεται εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να έχει μια ανεξάρτητη ε, πολιτική επιρροή. Έχει τη δυνατότητα με βάση την επιρροή που έχουν κερδίσει τα κράτη-μέλη, ε, με βάση τις προηγούμενες κατακτήσεις τους, όπως ε, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αφέλεις απέναντι στις πολυβεριανές διακηρύξεις ούτε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της πολιτικής για αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια πολιτική που ε, οδηγεί προς τη φτώχεια τον ε, πληθυσμό. Εμείς δεν πρέπει ούτε να μπούμε στον ουτιλιτερισμό, ούτε στον ε, κολεκτιβισμό. Όμως και πάλι βλέπουμε ότι ακολουθούμε και πάλι τα εμπάργκο, όπως προτείνει η Ουάσιγκτον. Δεν μπορούμε να είμαστε αλληλεγγύοι του Γκουαϊντό, χωρίς, ε, που δεν αντιπροσωπεύει τις ε, ελπίδες των Βενεζολάνων, ούτε μπορούμε να ε, ακολουθήσουμε τον Μαδούρο που δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών του και πάλι για άλλη μια φορά είμαστε απλοί παρατηρητές. Ευχαριστώ πολύ. Από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Τέρτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ακούμε τον είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνεται η εντύπωση ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα οφείλεται σε μια φυσική καταστροφή. Επίσης, ε, όταν ακούμε και τους σοσιαλιστές, το ίδιο συμβαίνει. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι αιτίε αυτή τη τεράστια τραγωδία ε, που έχουμε ενώπιόν μα. Οι αιτίε είναι το καθεστώ. Είναι ένα σοσιαλιστικό τσαβιστικό καθεστώ που προκάλεσε μιζέρια στην πιο πλούσια χώρα τη Αμερική. Το καθεστώ στη Βενεζουέλα ε, έχει ε, ξεκινήσει με επιχειρήση για να συλλάβει τα μέλη της Συνέλευση και το Χουέγο για να μην επανακλεγεί. Δηλαδή συνεχίζεται η καταστολή. Και αυτή είναι η αιτία. Ήδη τεκμηριώθηκε ότι έχουμε 6.800 εξοδικαστικές εκτελέσεις σε 14 μήνες από την αστυνομία στη Βενεζουέλα. 6.800 εκτελέσεις σε 14 μήνες. Χιλιάδες υπέστησαν βασανιστήρια και σεξουαλικές ενοχλήσεις. Ε, όμως ε, δεν ε, λαμβάνονται επιλεκτικές κυρώσεις κατά αυτού του καθεστώς που έχει προκαλέσει τρομερές καταστροφές σε ειρηνική περίοδο. Σε μία συνέντευξη που δόθηκε σήμερα είπε ο κύριος Μπρέλο ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν θέλει να φύγει ο Μαδούρα έχουμε πρόβλημα. Όχι ένα πρόβλημα. Έχουμε πολλά προβλήματα κύριε Μπορέλ. Γιατί οι τυρανοί δεν φεύγουν ποτέ εθελούσια. Οι Βενεζολάνοι φεύγουν εκδιωμένοι και πεθαίνουν και πεθαίνουν πεθαίνουν κατά χιλιάδες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει την αξιοπιστία της με μια ανήθικη ανοχή. Δηλαδή είμαστε παθητικοί και αυτό μας κάνει συνενοχούς όλους σε αυτή την τραγωδία. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την QNGL. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ιντόγια Βιλερουέβα Ρουίς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι ο λόγο που μετά από τόσο καιρό ε, ε, η αστίαση που έχει γίνει και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων στην Βενεζουέλα. Σε μια κατάσταση πόλωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, πολιτική του Τραμπ ε, δέχτηκε τον αυτονοκηρυγμένο Γκουαϊντό και μπορώ να σα πω ότι εδώ ε, πρέπει να αναγνωρίζουμε κράτη, όχι κυβερνήσει και η συνέπεια είναι η πολιτική κρίση συνεχίζεται και οξύνεται η κοινωνική κρίση λόγω των κυρώσεων. Η αναγνώριση του Γουαϊντό δεν χρησιμεύσει σε τίποτα και οι κυρώσει ε, κατά τη κυβέρνηση ζημιών του πληθυσμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να είναι διαμεσολαβητής έχουμε την ευκαιρία του χρόνου ε, να γίνουν ε, βουλευτικές εκλογές. Σας εργαστούμε για να γίνουν με εγγυήσει με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων χωρίς προηγούμενα μποϊκοτάζ για να ολοκληρώσουμε κλείσει αυτή η περίοδος αστάθειας και εξωτερικών ε, παρεμβάσεων και ε, απόπειρα πραξικοπημάτων που απλώς έχουν βλάψει τον ε, λαό της Βενεζουέλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Η συζήτηση για τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα έρχεται σε συνέχεια ψηφισμάτων που αναγνωρίζουν τον αχυράνθρωπο των ηνωμένων πολιτειών αμερικής γκουαϊδό σαν προσωρινό πρόεδρο ενάντια στον εκλεγμένο πρόεδρο μαδούρο. η στάση της ευρωπαϊκής ένωσης στηρίζει το πραξικοπηματικό σχέδιο των ηνωμένων πολιτειών της αμερικής κρατών μελών της ομάδας της λίμα και του οργανισμού αμερικανικών κρατών. η φτώχεια τα προβλήματα που πλήττουν το λαό της βενεζουέλας η αρνητική κατάσταση στην οικονομία πατάνε στο έδαφος της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η οποία επιδεινώνεται από τις υπεριαλιστικές κυρώσεις από την παρέμβαση ηνωμένων πολιτειών της αμερικής και ευρωπαϊκής ένωσης στις εσωτερικές της υποθέσεις. οι υποκριτικές ευαισθησίες σας για τους πρόσφυγες δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα γνώριμο εργαλείο εργαλείο διείσδυσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μονοπωλίων σε τρίτες χώρες ιδιαίτερα όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν κυβερνήσεις της προτίμησής ιδιαίτερα σε μια χώρα πλούσια σε κοιτάσματα φυσικού αερίου πετρελαίου πολύτιμων μετάλλων όπως είναι η βενεζουέλα εκδηλώνεται και με αυτόν τον τρόπο η κούρσα των ηνωμένων πολιτειών αμερικής και της ευρωπαϊκής ένωσης ενάντια στους διεθνείς ανταγωνιστές τους που έχουν συνάψει εδώ και χρόνια συμφωνίες συνεκμετάλλευσης. καταδικάζουμε τα πραξικοπηματικά σχέδια ηνωμένων πολιτειών αμερικής και ευρωπαϊκής ένωσης στη βενεζουέλα με στόχο την ανατροπή του εκλεγμένου προέδρου εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στο λαό της βενεζουέλας στους κομμουνιστές που μάχονται για τα λαϊκά συμφέροντα. ο λαός της βενεζουέλας είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταγιάννη για 1,5 λεπτό. 7.000 άτομα ε, έχουν να αντιμετωπίσουν δίκε ε, και στην Βενεζουέλα έχουμε πάρα πολλού ε, διοκόμενου Από το 12 έχουν συλληφθεί πάρα πολλέ γυναίκε για πολιτικού λόγου. Η έκθεση τη κυρία Μπαρσελέ λέει ότι στην Βενεζουέλα έχουν δολοφονηθεί περίπου 5.000 άτομα το 2018 1.500 τόσα ε, μέχρι το Μάρτι του 2019. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία. Αυτοί είναι κύριε οι θαραλέοι κομμουνιστές που θέλετε εσείς να υπερασπιστήσετε. Εκατομμύρια ή χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να εγκαταλείψουν την Βενεζουέλα. Πάρα πολλοί δολοφονούνται. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει και διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών. Η ελευθερία της έκφρασης δεν υπάρχει. Εξαφανίζονται οι εφημερίδες. Ε, πολλοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε στο κινητό τηλέφωνο, ούτε στο ίντερνετ. Έχουμε ένοπλε δυνάμει που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια, δεν έχουμε φάρμακα, ε, αυξάνεται, αυξάνονται οι ασθένειε, η ελεονοσία, η φηματίωση Άρα δηλαδή, ε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, θα πρέπει να ερωτηθεί κανείς κατά πόσον η κατάσταση στην Βενεζουέλα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια. Μα δεν ξέρουμε καν πού φτάνουν αυτά τα, που φτάνει αυτή η βοήθεια. Το καθεστώ του Μαντούρο φιλτράρει και αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, υπάρχουν προβλήματα στη δημοκρατία, κύριε Μπορέλ. Πρέπει να έχει κανεί περισσότερο θάρρο. Μέχρι σήμερα οι ενωσιακοί θεσμοί, εκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είχαν το θάρρο να στείλουν στο σπίτι του τον κύριο Μαδούρο. Να είναι άκαμπτη και κατηγορηματική έναντι ενό ανθρώπου που έχει κατακρεουργήσει το το λαό του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και εσείς και οι ενωσιακοί θεσμοί να δείξουν κάποιο θάρρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Μαρία Μανουέλ Τάο Μαρκές ε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πατακπρόσωπε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση σήμερα. Αν δεν αλλάξει τίποτα, προβλέπεται ο ρυθμός των προσφύγων και των μεταναστών στη Βενεζουέλα από 4,5 εκατομμύρια θα φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια το Δεκέμβριο του 2020. Αυτή η κρίση πλήττει την ε, περιοχή και τις γειτονικές χώρες και ιδίως την Κολομβία μέχρι και την Ευρώπη. Μάλιστα στην ε, Μαδέρα, στην Πορτογαλία, σε αυτό το μικρό νησί το 2018 ήδη είχαν ε, φτάσει και είχαν ενταχθεί περίπου 4.000 μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση, είναι και αυτή που στηρίζεται λιγότερο οικονομικά. Μόλις το 48% των ε, χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δωρητές υλοποιήθηκαν το 2019. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει το έργο τη σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οικονομικέ δεσμεύσει και επίση να αξιολογηθεί ο αντίκτυπο των οικονομικών κυρώσεων μελετώντα ενδεχόμενε εναλλακτικέ με δημιουργικότητα όπω ε, αυτή που υπεράσπισε ο ύπατο εκπρόσωπο ε, προλίγου ένα πρόγραμμα όπω το Oil for Food. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χορδικάνιας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Βενεζουέλα βιώνει μια πραγματική κατάσταση επίγουσα έκτακτη ανθρωπιστική ανάγκη. 4,5 εκατομμύρια εξορίστηκαν και τελικά μπορούν να φτάσουν τα 6 εκατομμύρια το 2020. 5.000 καθημερινά εγκαταλείπουν τη χώρα του και ε, δεν έχουμε κάποιο πόλεμο εκεί, ούτε κάποια ξαφνική φυσική καταστροφή. Έχει έναν υπεύθυνο που λέγεται Νικολάς Μαδούρο και ένα καθεστώς που τον προστατεύει. Και μπροστά σε αυτήν την κατάσταση τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι πολύ απλό, όπως να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Και λέω τόσο απλό, γιατί όλα τα υπόλοιπα απλώς διονύσουν την κατάσταση. Και οι πολίτε στη Βενεζουέλα πρέπει να ακούσουν μια ξεκάθαρη φωνή από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο, που να του πει ότι θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, γιατί έχουμε εξοδικαστικές εκτελέσει στη Βενεζουέλα, διώκονται η πολιτική, υπάρχουν πολιτικοί κρατουμένοι και δολοφονούνται οι ηθαγενικές κοινότητες. Ξέρετε τι συμβαίνει. Κάποιοι ε, εδώ κοιτάνε από την άλλη πλευρά όμως ε, οι περισσότεροι θα κοιτάξουμε στα μάτια του δικτάτορα και θα του πούμε θα τελειώσουμε μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σιλβία Σερντόνε για ένα λεπτό. Για πολλωστή φορά όσον αφορά την ε, Βενεζουέλα βλέπουμε πόσο άχρηστη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Μαδούρο η Ευρώπη είχε απογοητευτική στάση. Δεν υπήρξε σαφής επίθεση απέναντι στο κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο είχε εφεύρει ο Τσάβες και μετά υιοθέτησε και ο Μαδούρο. Είναι ένα μοντέλο το οποίο στη Βενεζουέλα σε μια πλούσια χώρα σε πετρέλαιο έφερε την πείνα. Ε, περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού αποφάσισε μεταναστεύσει, να φύγει, ε, άδεια τα μαγαζιά, ε, πάρα πολλές ασθένειες, λείπουν τα φάρμακα. Ε, βλέπουμε λοιπόν μια διάχυτη κατάσταση και αναγκάζονται να φάνε άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ποιο είναι το σοσιαλιστικό μοντέλο. Τι ακριβώς είναι ο υπαρκτός σοσιαλισμός, τι είναι ο κομμουνισμός. Είναι κάτι το οποίο φέρνει μόνο φτώχεια και θάνατο. Αυτό είναι ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός και ε, γι' αυτό το λόγο ε, δεν υπάρχει ελευθερία τύπου, ε, δεν υπάρχουν εκλογές. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Τόμας Πιότρο Πορέμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στην Λατινική Αμερική. Επομένω, ε, όλοι θα έπρεπε να ζουν με ευημερία και να επιτυχαίνουν τα όνειρά του. Δυστυχώ όμω δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ήδη έχουμε συζητήσει για τη Βενεζουέλα και στο παρελθόν και είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εκατομμύρια έχουν φύγει από τη χώρα. Έχουν υπάρξει εξοδικαστικές ε, δολοφονίες. Εκατοντάδες μάλιστα. Επομένω, ε, θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προ αυτή τη χώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανεχθεί πια τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Και καλό τον κύριο Μπορέλ στα επόμενα χρόνια να απευθύνουμε αυτή την έκκληση για να διευρυνθούν οι κυρώσεις ε, προς ε, το καθεστώς και να απευθύνουμε έκκληση για μια ισχυρή δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Εκτός και αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μια ισχυρή κοινή νέα φωνή, δεν θα καταφέρουμε να ε, αλλάξουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κύριε Περέρα. Ευχαριστώ αυτό το κοινοβούλιο ε, συζητά περιοδικά το θέμα της ε, δημοκρατίας, της βολιβερινής δημοκρατίας της ε, Βενεζουέλας. Όμως εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για παρέμβαση αφού έγιναν ε, πολλές απόπειρες πραξικοκλήματος, τρομοκρατίας, σαμποτάζ και όλο και πιο σοβαρές κυρώσεις είναι υποκριτικό να αναφερόμαστε σε μεταναστευτικά φαινόμενα χειρογόντας τις αντιμεκενικές συνθήκες ή η ειρήνη, η απασχόληση, η η κοινωνικη προστασια υγειονομική περίθλιψη, καταπολέμηση της φτώχεια μια πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξης είναι ουσιαστικοί παράγοντες ε, για ε, την προστασία του βιωτικού επίπεδου. Διαφορετικά έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Τα συμφέροντα του λαού της Βενεζουέλας και της ε, πορτογαλικής κοινότητας στη χώρα αυτή δεν είναι συμβατά με αυτή την αστάθεια. Εμεί δεν συμφωνούμε με την χρησιμοποίηση των δεινών του λαού και απαιτούμε να αρθούν όλες οι κυρώσεις που ζημιώνουν το λαό της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαγός για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κάνω ακούω μια κουβέντα η οποία κατά την άποψή μου είναι άκρο υποκριτική. Και είναι υποκριτική γιατί σύμφωνα με όλα τα δεδομένα δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή ένωση για να σταματήσει αυτό που συμβαίνει στη βενεζουέλα όπω δεν μπορούσε να το σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουν ξαναγίνει τέτοιε συζητήσει όπω δεν έχει μπορέσει να το σταματήσει και σε άλλα κράτη στα οποία αποδεδειγμένα υπάρχει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. οπότε να δούμε και να συμφωνήσουμε σε τι στο ότι το καθεστώ τη βενεζουέλα έχει δημιουργήσει μια απαράδεκτη στάση και απαράδεκτη κατάσταση για του κατοίκου τη χώρα βεβαίω. Ποιο καθεστώ είναι εκεί πέρα όμω, μην ξεχνάμε ότι είναι το κομμουνιστικό καθεστώ. Είναι το κομμουνιστικό καθεστώ που όπου έχει επικρατήσει, όπου έχει πάρει τα ενία στα χέρια του, έχει ισοπεδώσει πραγματικά του ανθρώπου. Έχει ισοπεδώσει του ίδιου του πολίτε των χωρών του. Άρα, να ξεκινήσουμε από εκεί και να δούμε και τι άλλο γίνεται, να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να σταματήσει κάτι τέτοιο. Αποδεικνύεται πω όχι. Και απλά κάνουμε κουβέντε απλά για να τι κάνουμε. Συζητάμε για να συζητάμε. Και πώ θα μπορούσε άλλωστε να επιβληθεί η γνώμη και η άποψη τη ευρωπαϊκής Ένωση στη βενεζουέλα ή σε κράτη που είναι τόσο πολύ μακριά από εμάς όταν εδώ δίπλα μας στα σύνορα της ευρώπης στα σύνορα με την πατρίδα μου στην ελλάδα η τουρκία κάνει ό,τι θέλει ένα στιγνός δικτάτορας κατά την άποψή μου ο ερντογάν κάνει αυτό που πραγματικά θέλει εκεί έχει ανοίξει τα σύνορα και περνάει τους λαθρομετανάστες σοριδών στην ευρωπαϊκή ένωση απειλεί και συνεχώς κερδίζει. κάνει ό,τι θέλει παίρνει μάλιστα και παχυλά κονδύλια από την ευρώπη προκειμένου να κάνει όλα αυτά. κοιτάξτε λοιπόν πώς θα σταματήσετε όλους αυτούς που είναι εδώ δίπλα στη γειτονιά μας και μετά σιγά σιγά μπορούμε να σταματήσουμε και τους άλλους που είναι πιο μακριά από εμάς. Ευχαριστώ. Ο Παύλο uh, Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι απορρίπτω κατηγορηματικά όλες τις δηλώσεις της κυρίας Περέιρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας που ε, προσπαθεί να παρουσιάσει και να υπερασπίσει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς όπως του Μαδούρο. Είναι ντροπή να υπάρχουν βουλευτές εδώ σε αυτό το νοικό που υπερασπίζουν τις πολιτικές ε, του Μαδούρου που οδήγησαν στην μεγαλύτερη μετατόπιση ε, πληθυσμού στην Αμερικανική Ήπειρο στην ιστορία του και τώρα ε, ε, πάει ε, μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσουν τα 6,5 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. πολλοί έχουν πάει στην Κολομβία, στο Περού, στη Βραζιλία, στη Χιλή. Ξέρω ότι είναι σε απελπιστική κατάσταση οι άνθρωποι αυτοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και οφείλει να κάνει περισσότερα και τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνε για να θέσουν τέλο στο καθεστώ του Μαδούρου και να αποκαταστήσουν τη δημοκρατική νομιμότητα στη Βενεζουέλα προκειμένου να ευμερεύσει εκ νέου ο λαό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίτσουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε είπατε 4,5 εκατομμύρια πολίτε έχουν ήδη φύγει από τη Βενεζουέλα και μέχρι τα τέλη τη επόμενη χρονιά αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια αυτό ο αριθμό. Ε, πρόκειται σαφώ για το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από μία χώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτό συνοδεύεται και από πολύ χαμηλή, χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης από την διεθνή κοινότητα. 320 εκατομμύρια έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστική βοήθεια το 2016. Όμω θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια και στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία και στο Περού. Αυτέ οι χώρε έχουν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ε, προ τη Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά του πρόσφυγε. Το 80% των προσφύγων πηγαίνει στι γειτονικέ χώρε. Ε, στηρίζω την προσέγγιση της υπατησαρμοστίας. Δεν θα πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν το τίμημα και τις κυρώσεις. Η κρίση με τη Βενεζουέλα θα πρέπει να λήξει μέσω διαπραγματεύσεων και μέσω δίκαιων εκλογών με την παρουσία διεθνών ε, παρατηρητών. Μόνο έτσι μπορούν οι ίδιοι πολίτες να αποφασίσουν ποιο θέλουν να είναι το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ραφαέλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Έξι μήνε έχουν περάσει από τότε που ήρθα εδώ για πρώτη φορά. Και πάλι συζητούσαμε για τη Βενεζουέλα τότε. Τα νούμερα μιλούν από μόνα του. 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα. 1,5 εκατομμύριο έχει πάει στην Κολομβία. Χιλιάδε Βενεζουελάνοι ε, βρίσκονται στα, ε, στις εκτάσεις ε, στην Καραϊβική της Ολλανδίας τι συμβαίνει το τελευταίο εξάμεινο. Δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σίγουρα. Και στην Αρούμπα και στα υπόλοιπα αυτά ολλανδικά νησιά ε, των αντιλών δεν υπάρχει κάποια βελτίωση. Πρέπει να στηρίξουμε καλύτερα τις ε, ευρωπαϊκές πλέον απομακρυσμένες περιοχές μας. Και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το ε, Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο ε, Κοινωνικής Ένταξης και ασύλου και να τους ε, βοηθήσουμε και με τις υποβολές ε, των ετοιμάτων ασύλου. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Ο κύριος Μπορέλ είναι Ισπανός ε, και έρχεται από μια χώρα που κατανοεί τα προβλήματα της ε, Λατινικής Αμερικής. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύριος Μπορέλ ε, θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Όμως, ας μην είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Οι δικτατορίες ε, δεν αναστέλλονται από τη μία μέρα στην άλλη. Οι αρχές ε, στη Βενεζουέλα στηρίζονται μόνο στην καταστολή, στην σωματική βία, άρα δηλαδή μόνο πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι δηλαδή μόνο διπλωματία, αλλά πραγματική πίεση μπορούν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους Βενεζουάλους για να αποφασίσουν ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο αγέτης ε, της χώρας τους. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν 4,5 εκατομμυρία άτομα εγκαταλείπουν τη χώρα του, αν οι γονεί δεν μπορούν να δώσουν τροφή στα παιδιά του, ε, αν ο ετήσιο πληθωρισμό είναι περίπου 10.000%, τότε μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι του χρόνου ο αριθμός των Βερζολάνων ε, μεταναστών θα υπερβεί τους Σύρους ε, πρόσφυγες με 6 εκατομμύρια το 2021. Έχουμε περίπου 2,5 ε, εκατομμύρια Βενεζολάνου στην Κολομβία, μια χώρα που κράτησε πολιτική ανοιχτή πόρτα και που τώρα πληρώνει πολύ ακριβά τι ε, συνέπειε ε, τη υποδοχή τόσο μεγάλου ρυθμών ανθρώπων. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν τι ανθρωπιστικέ ανάγκε σε 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια δολάρια μόνο για να δοθούν ε, οι βασικές ε, υπηρεσίες ε, στους μετανάστες και για να υποστηριχθούν οι χώρες υποδοχής. Η πραγματικότητα είναι αν και πολλοί εκφράσουν αλληλεγγύη, τελικά πολύ λίγοι συνεισφέρουν. Γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια για να υποστηρίξει αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους και να ζητήσει από τις ΥΠΑ να θεωρήσουν την πολιτική κυρώσεων που παραλύουν ακόμη περισσότερο μια οικονομία που καταραίει. Ξέρω ότι η Βενεζουέλα είναι πολύ πιο μακριά από τη Συρία και πολλοί πιστεύουν ότι δεν μας πλήττει άμεσα αυτή η κρίση. Όμως πρέπει να δείξουμε στους φίλους μας στη Λατινική Αμερική ότι ε, όταν μας χρειάζονται είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κοβάτσεφ ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπορέλ. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια Βενεζουάλων έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την αρχή της κρίσης. Η κρίση αυτή προέκυψε λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τσάβες και του Μαδούρο και σε αντίθεση με άλλα μεταναστευτικά ρεύματα που υπήρξαν κατά διάρκεια όλων αυτών των ετών. Αυτό το μεταναστευτικό κύμα προέκυψε λόγω ενός ε, καθεστώτος ε, που είναι ιδιαίτερα διεφθαρμένο. Έχουμε μία από τις πιο πλούσιες ε, χώρες του κόσμου και όσοι από εμάς ζήσαμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα κατά το παρελθόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζει κάτω από κομμουνισμό. Τότε δεν είχαμε να φάμε, ήταν κλειστά τα σύνορα, υπήρχε έλλειψη πολλών αγαθών. Ε, θυσιάσαμε λοιπόν πάρα πολλά και κατορθώσαμε να ανατρέψουμε τα παλαιότερα τα πρώην καθεστώτα. Γι' αυτό το λόγο εμείς τώρα προσφέρουμε την υποστήριξή μας στους Βενεζουελάνους. Κύριε Μπορέλ, ας ε, καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειαζόμαστε ανώθευτες δημοκρατικές